και τα εγκεκριμένα κείμενα τα έχετε λάβει. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, θεωρούμε ότι τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται ούτω. Οι αρμόδιε αρχέ ε, του Ηνωμένου Βασιλείου μου ανακοίνωσαν ότι η κυρία Ελίζα Βεθλίντ θα αντικατασταθεί από τώρα, τον, από 6 Φεβρουαρίου του 2012, από τον κύριο Φίλ Μπενιόν. Τον καλωσορίζω. Είναι εδώ ο κύριο Μπενιόν. Πού είναι? Herr Μπενιόν. herzlich willkommen. Σας καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung ich erinnere daran dass jedes mitglied mit vollen rechten an den sitzungen des parlaments und seiner organe teilnimmt solange sein mandat nicht geprüft